οι αλλαγές αυτές εγκεκριμένες. Και τώρα να σας πω ποιες είναι οι προθεσμίες για την υποβολή τροπολογιών για τον προϋπολογισμό του 2015. Για τις επιτροπές και για τα μέλη τα οποία βασίζονται στον κανονισμό των 40 βουλευτών, η προθεσμία είναι η 5η 4 Σεπτεμβρίου 2014 στις 12 το μεσημέρι. Οι ομάδες ή τουλάχιστον 40 βουλευτές. 4 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι για τις ομάδες 11 Σεπτεμβρίου 2014 στις 12 το μεσημέρι και πάλι η προθεσμία. Οι αρμόδιες επιτροπές υπέβαλαν ε, διορθωτικά για έξι κείμενα σύμφωνα με τον κανόνα 231 παραγραφός 4.